Καλώς ε, ήρθατε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας αρχίσουμε την διαδικασία ε, ψηφοφορίας. Υπάρχουν πολλά θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξή μας σήμερα. Υπάρχει πρώτα ένα διαδικαστικό του κυρίου Καρύμ. Κύριε Πρόεδρε, η εφημερίδα Φιγκαρό λέει σήμερα ότι ένας δημοσιογράφος όχι μόνο εισήλθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ένα ψεύτικο όπλο, αλλά μπόρεσε μάλιστα να πλησιάσει πάρα πολύ τον πρίγκιπα Κάρολο, διάδοχο του Βρετανικού θρόνου με τις ανησυχίες που έχουμε για την ασφάλεια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε σήμερα ότι λαμβάνετε πολύ σοβαρά υπόψη το θέμα αυτό και ότι αυτή η επανεξέταση που υποτίθεται ότι γίνεται εν κρυπτό και παραβίστο από το ε, Προεδρείο του Κοινοβουλίου θα οδηγήσει σε μια σε βάθος ε, μεταρρύθμιση των θεμάτων ασφάλειας. Thank you, Mr. Karim. I can ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Σας διαβεβαιώ ότι το θέμα αυτό λαμβάνεται πραγματικά πολύ σοβαρά υπόψη και από τις πληροφορίες που γνωρίζω συζητείτε στην διάσκεψη Προέδρων Πολιτικών Ομάδων. Να είστε λοιπόν βέβαιος ότι το ε, Κοινοβούλιο αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το σοβαρό θέμα. Ας αρχίσουμε τώρα. Το θέμα το κείμενο μάλλον για τον νόμο τύπου στην Ουγγαρία θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Προτείνω λοιπόν να αναβληθεί η σχετική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 177 παράγραφος 4 του κανονισμού. Η απόφαση για περαιτέρω δράση για το θέμα αυτό καθώς και οι νέες προθεσμίες θα οριστούν στην διάσκεψη των Προέδρων Πολιτικών Ομάδων την 5η 3 Μαρτίου. Επιθυμεί κανείς να λάβει τον λόγο υπέρ της προτάσεως αυτής. Ουδής είναι υπέρ. Ουδής επιθυμεί να μιλήσει υπέρ. Επιθυμεί κανείς να μιλήσει κατά της προτάσεως αυτής. Η κυρία. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω μετά πράγματι από τις τελευταίες εξέλιξεις που τέθηκαν και υπόψη ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι όμως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να αναβάλουμε την ψηφοφορία για το ψήφισμα το οποίο πρέπει να τροποποιηθεί για να αποδίδει τις νέες αυτές εξελίξεις. Σε ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Αυτό ήταν λοιπόν μια τοποθέτηση υπέρ. Ποιος επιθυμεί να τοποθετηθεί κατά. Ουδής. Τότε ας ψηφίσουμε ψήφι υπέρ της αναβολής. Κατά αποχές εγκρίνεται η αναβολή, άρα το ε, θέμα αυτό αναβάλλεται. Η ψηφοφορία μάλλον αναβάλλεται. Ακολουθεί η ψηφοφορία για την έκθεση του κ. Ζάλμπα Μπιντεγκάιν για θέματα ε, συμφωνίας τροπολογία πρώτα 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροποποιημένες τώρα ε, τροπολογίες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το νομοθετικό περιεχόμενο ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει λοιπόν τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ακολουθεί το επόμενο θέμα που είναι έκθεση του κυρίου Καλφίν για χορήγηση εγγύηση τη Ευρωπαϊκή Ενώση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγκυρίσει για σχέδια εκτό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Στο, στο σύνολό του το κείμενο, αλλά υπάρχει πρώτα μία προφορική τροπολογία. Εσείς κύριε Καλφίν. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, εν ώψη των πρόσφατων εξελίξεων στην ε, Βόρεια Αφρική και εν ώψη των επιπτώσεων των εξελίξεων αυτών καθώς και των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προτείνω μια προφορική τροπολογία με ορισμένους αριθμούς στην έκθεση. Η τροπολογία έχει ως εξής για το παράρτημα 1 για το Β γειτονία και θα πρέπει να είναι 30 εκατομμύρια για τις χώρες Μεσογείου 9.700.000. Θα χρειαστεί να διορθωθούν οι αριθμοί στο, στο άρθρο 2 παράγραφος 1. Το σωστό θα είναι 29.567.000. Σας ευχαριστώ κύριε Καλφίν. Υπάρχουν ε, αντιρρήσεις. Δεν βλέπω να υπάρχουν ε, ενστάσεις τίθεται σε, τροπολογία, σε ψηφοφορία η τροπολογία υπαριθμών 1 αρχίζει ονομαστική ψηφοφορία πέρας εγκρίθηκε τροπολογία 5 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία υπαριθμών 2, ονομαστική ψηφοφορία, αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 3, πάλι ονομαστική ψηφοφορία, αρχίζει. Εάν κάποιος έχει, αντιμετωπίζει προβλήματα με το μηχάνημα, θα στείλουμε μέσω τεχνικό. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τώρα όσοι τροποποιήθη, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, νομοθετικού περιεχομένου ψήφισμα, ονομαστική ψηφοφορία, αρχίζει. Πέρας. εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια στον κύριο εισηγητή. Ακολουθεί η έκθεση Στέρντι, Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημοκρατίας της Κορέας. Βλέπω ότι ο εισηγητής ζητεί να λάβει το λόγο. Εγώ επιθυμώ να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και τους κοιόδης συγητές για την ε, συνεργασία. Πρόκειται για μια πραγματικά ρηξικέντευτη συμφωνία εμπορικών συναλλαγών που δίνει μια μεγάλη ευκαιρία έχει τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μάλλον τη μεγάλη ευκαιρία να υποστηρίξει ε, ένα σύνολο ιδεών που θα είναι πραγματικά πολύ σημαντικές για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Θέτω λοιπόν αυτή την ε, απίθανη συμφωνία σε ονομαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια κύριε Στέρντι. Ακολουθεί ψηφοφορία επί 7 προτάσεων ψηφισμάτων και την κατάσταση στην Αίγυπτο. Αρχίζουμε με την παράγραφο 9 που προβλέπει χωριστή, δύο ψηφοριστικά τμήματα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Παράγραφος 10, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος ονομαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 11. Πρώτο μέρος, ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 15. Πάλι το πρώτο μέρος, το πρώτο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Πέρας. εγκρίνεται και αυτό. Το δεύτερο μέρος, το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε στο σύνολο του ψηφίσματος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφοφορία επί τριών ψηφισμάτων για την στατική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη. Έχει αποσυρθεί η τροπολογία υπαριθμών 1. Ψηφίζουμε λοιπόν στο σύνολό του το ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψήφι, ε, ε, αρχίζει μάλλον η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με σαφή πλειοψηφία. Έχουμε τώρα έξι προτάσεις ψηφισμάτων για το κράτος δικαίου στην Ρωσία. Το σύνολο του λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ακολουθεί ψηφοφορία της Επιτροπής της Επιτροπής Αναπτύξεως για την Ενεργειακή Στρατηγική της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αρχίζουμε με την παράγραφο 2. Ζητείται ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αυτό εδώ καλά θέλετε λοιπόν να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει πέρας εγκρίθηκε Τώρα έχουμε την τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ κατά χέσα. νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε και πάλι ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας εγκρίθηκε περνάμε τώρα στην τροπολογία υπαριθμών 2 ποιοι είναι υπέρ κατά χέσα. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην παράγραφο 7, χωριστή ψηφοφορία, πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε και πάλι ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος υπαριθμών 10 και πάλι χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά και πάλι άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Περνάμε στο δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην τροπολογία υπαριθμών 3. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος υπαριθμών 12 και πάλι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε και πάλι ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται Τώρα περνάμε στην αιτιολογική σκέψη Α, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη γ τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ε, ψηφίζουμε για το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια. Το επόμενο θέμα έχουμε έξι προτάσεις ψηφίσματος για την Ευρώπη 2020. Αρχίζουμε με την παράγραφο 3 χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πρόκειται για ονομαστική ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας τη ψηφοφορία. Και εγκρίθηκε. Τώρα έχουμε την τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ο κύριος Μπούλμαν έχει προφορική τροπολογία. Έχετε το λόγο κύριε Μπούλμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας επιθυμώ να υποβάλω προφορική τροπολογία για να περιληφθεί το θέμα της ισότητας των φύλων. Διαβάζω το κείμενο στα αγγλικά. Νέα παράγραφος 10α επιμένει ότι η ισότητα των φύλων είναι στόχος κλειδί για να επιτευχθεί μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης 2020 με πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και με πλήρη συμμετοχή γυναικών εργαζομένων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Επίσης, να δημιουργηθεί ατζέντα για να εξαλειφθεί το, το χάσμα αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ευχαριστώ. Υπάρχει κανείς κατά. Ψηφίζουμε λοιπόν για την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, παράγραφο 12 και πάλι σε δύο μέρη. Για το πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ε, ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Ναι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13 και πάλι σε δύο τμήματα. Ονομαστική ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Επίσης εγκρίθηκε παράγραφος 20. Πρώτο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Παράγραφος 21. Πρώτο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 23. Πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται σαφώς δεύτερο τμήμα αρχίζει η ψηφοφορία αρχίζει η ψηφοφορία αχ κάποια σύγχυση άρχισε η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας τώρα εγκρίνεται τώρα έχουμε την ε, τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 26. Ε, Ποιοι είναι υπέρ, ε, εγκρίνεται. Τώρα ψηφίσουμε για το ψήφισμα στο σύνολό του. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Το επόμενο θέμα είναι η πρόταση ψηφίσματος από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών για την πολιτική των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης. Αρχίζουμε με την παράγραφο 4, ονομαστική ψηφοφορία, άρχετη ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται με σαφή πλειοψηφία. Παράγραφος 7 Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Ποιοι είναι ε, υπέρ, εγκρίνεται. 19 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές. Διαδικαστικό. Είμαι υποχρεωμένος να διακόψω τη διαδικασία διότι δεν λειτουργεί το μηχάνημά μου κύριε Πρόεδρε. Θα σα στείλουμε αμέσω τον τεχνικό, απαντά ο πρόεδρο. Τώρα θα ψηφίσουμε για το ψήφισμα στο σύνολό του. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε για την έκθεση της κυρίας Μπέρενς για τις κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόληση των κρατών μελών, νομοθετικό ψήφισμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Είχατε όλοι χρόνο να ψηφίσετε. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται σαφώς. Το επόμενο θέμα είναι η ψηφοφορία για έξι προτάσεις ψηφίσματος για τις αυξανόμενες ε, τιμές προφήμα, τροφίμων, ονομαστική ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε τροπολογία 6, ονομαστική ψηφοφορία, αρχιετή ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. και πάλι απορρίφθηκε. Τροπολογία 8, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Και για τρίτη φορά απορρίφθηκε τροπολογία. Τώρα παράγραφος 5 σε δύο τμήματα, χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα έχουμε την... Θέλετε έλεγχο. Ας ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 5. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Είχατε δίκιο. Τώρα περνάμε στην τροπολογία 9. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Έχουμε την παράγραφο 6 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Παράγραφος 10, σε δύο τμήματα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, μπορούμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά αν θέλετε. Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά σε ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε σαφώς. Σας παρακαλώ να σηκώνετε καλά τα χέρια την επόμενη φορά. Παράγραφος 13 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Έχουμε τώρα την τροπολογία 11, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τώρα μετά την έχουμε την ε, τροπολογία 10, ανομαστική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Παράγραφος 21. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε παράγραφος 23 σε τρία τμήματα πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψηφίζουμε για το τρίτο τμήμα Πέρας της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. Τώρα παράγραφος 27 και πάλι χωριστή ψηφοφορία έχουμε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Τώρα έχουμε την τροπολογία 7, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με τρεις ψήφους επιπλέον. Σε αυτήν την περίπτωση περνάμε στην τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχέσα, απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Ε, τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Δεν είναι σαφές. Ίσως είσαστε κουρασμένοι. Ας, προ... ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 4 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίφθηκε αιτιολογική σκέψη Δέλτα, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε για το ψήφισμα στο σύνολό του, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά σχετικά με τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Χρειάστηκαν 28 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Τώρα θα έχουμε επεξηγήσεις ψήφων.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 Θα ακούσουμε τώρα τις ε, αιτιολογήσεις ψήφου. Πρώτα για την έκθεση Bidegain. Πρώτος ο κ. Μικολάσικ.